να μην εκφραστεί για μια ε, κατεξοδότηση πράξη και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών βάσει το 156 μου το ανακοίνωσε. Μου ανακοίνωσε ότι στη διάσκεψη των Προέδρων δεν υπήρξε καμία αντίρρηση για αυτήν την ενέργεια. Να μην έχει αντίρρηση σε μια κατεξοδότηση πράξη. Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση από πλευρά πολιτική ομάδα 24 ε, ε, ωρών ή από τουλάχιστον 40 βουλευτές τότε θα θεωρεί ότι εγκρίθηκε. Τη σύσταση θα τη βρείτε στο site της Ολομέλειας. Σήμερα μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή καλύτερα την πρόεδρο του Συμβουλίου